συνέντευξη των ε, Προέδρων στις 5 Μαρτίου ενέκρινε σύμφωνα με το άρθρο 149 του κανονισμού το τελικό σχέδιο μερίσιας διάταξης. Το έχετε λάβει. Για σήμερα δεν έχει ζητηθεί καμία τροποποίηση ούτε για αύριο, Τρίτη. Για την Τετάρτη υπάρχει ένα αίτημα από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ε, υπάρχει μια συζήτηση δήλωση της Επιτροπής για την άνοδο του αντισημιτισμού, την Ισλαμοφοβία και το βίο εξτρεμισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ΕΛΚ ζητεί να υπάρξει και ψήφισμα, το οποίο θα ψηφιστεί στη δεύτερη σύνοδο του Απριλίου. Για να αιτιολογήσει το αίτημα, το λόγο έχει η κυρία Μέτσολα. Ευχαριστώ να γίνει αργότερα στην εβδομάδα συζήτηση για την έξαρση του αντισημιτισμού και του, της ξενοφοβίας τα από και μάλιστα να συνταχθεί και ψήφισμα για την, για την Ολομέλεια του Απριλίου. Διαφωνεί κανείς. Κυρία Χόλμαγερ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, αυτό το θέμα του αντισημιτισμού και του βίαιου εξτρεμισμού θέλουμε να συνοδευτεί από ψήφισμα για να στείλουμε ένα κοινό μήνυμα. Χωρίς όμως λεπτομέρειες, ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλουμε να εκφράσουμε αυτό που ε, εκφράζουμε και στις ε, εκθέσεις ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα που υποστηρίζουν και οι άλλες πολιτικές ομάδες, οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες, οι γκούε, οι φιλελεύθεροι. Δεν χρειάζεται να σας εξηγήσω για ποιο λόγο. Σχεδόν κάθε εβδομάδα έχουμε διάφορες επιθέσεις και έκτροπα. Και θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα με το ψήφισμα ότι το Κοινοβούλιο είναι ενωμένο, είναι συντεταγμένο και θέλει να ακουστεί ισχυρά η φωνή του την Επιτροπή μας Ελευθεριών έχουμε προβλέψει να κάνουμε ακρόαση και επί της ουσίας να αναλάβουμε πρωτοβουλίες. Οπότε αυτό το ψήφισμα παρακαλώ να το εκλάβετε ως μήνυμα ως ένα ηχηρό μήνυμα ε, διακομματικό που να συμφωνήσουν στο ψήφισμα όλες οι ομάδες κατά του αντισημιτισμού και ε, του εξτρεμισμού ε, του βίαιου. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό ήταν υπέρ. Ποιο θέλει να μιλήσει κατά, ε, κυρία Ζίπελ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, εάν ε, είμαι καλά πληροφορημένη, ήδη στη διάσκεψη των Προέδρων είχε τεθεί αυτό το αίτημα, η συζήτηση για τον αντισημιτισμό και τα λοιπά να συνδεθεί με ψήφισμα. Και στη διάσκεψη των Προέδρων αυτό απερίφθη. Δεν αμφισβητεί κανείς ότι αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ λεπτό και χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, ειδικά του αντισημιτισμού σε κάποια από τα κράτη-μέλη μας. Αλλά θέλουμε να το κάνουμε με διαφορετική σειρά εμείς. Το μήνυμα ε, εκπέμπεται ήδη από τη συζήτηση που έχουμε αυτή την εβδομάδα. Και μετά θέλουμε, σε μια κρόαση που ήδη έχει αποφασιστεί, να ασχοληθούμε συστηματικά, όχι μόνο με την ιστορική εξέλιξη του αντισημιτισμού και της Ισλαμοφοβίας ε, και όχι μόνο με τα σημερινά φαινόμενα, αλλά και με τα μέτρα και τα βήματα που μπορούμε να κάνουμε εμείς ε, Λέω στην ακρόαση λοιπόν σε βάθος να το συζητήσουμε και ένα ευρύτερο στη συνέχεια ψήφισμα να περιλαμβάνει όλα τα αποτελέσματα. Επαναλαμβάνω, δεν είμαστε κατά του ψηφίσματος, αλλά όχι τώρα. Χρονικά θα πρέπει να προηγηθεί η ακρόαση και να ακολουθήσει το ψήφισμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ψηφίζουμε. Ποιο είναι υπέρ του αιτήματο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο, παρακαλώ. Κατά. Αποχέ. Χρειάζεται μάλλον ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Επαναλαμβάνω, ψηφίσατε όλοι. Κοιτάξτε, πρώτο σηκώσατε χέρι και τελευταίος ψηφίζετε ηλεκτρονικά. Αλλά επειδή είμαι πολύ επίκης και γενναιόδωρος, πέρασε ψηφοφόρες. 152. Ισοψηφία. 152-152. Αν δεν σας είχα δώσει κύριε Μπουτικόφερ την ευκαιρία να ψηφίσετε, ποιος ξέρει τι θα έβγαινε. Απορρίπτεται λοιπόν το αίτημα αυτό και λυπάμαι πάρα πολύ. Προχωρούμε. Πέμπτη. Την Πέμπτη. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ζητεί Ω δεύτερο σημείο στην ημερήσια διάταξη, δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ενδεχόμενο κύμα ε, ε, μεταναστών στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της ε, πρόσφατης προέλασης του Ισλαμικού κράτους στη Λιβύη, χωρίς ψήφισμα. Η κυρία Χολμάιρε έχει το λόγο για να εξηγήσει το αίτημα αυτό του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Με μεγάλη ανησυχία όλες οι χώρες της Μεσογείου παρατηρούν την κατάσταση στη Λιβύη και για το λόγο αυτό θα επιθυμούσαμε παρακαλώ η κυρία Μογκερίνη να έρθει στο Κοινοβούλιο και να ε, λογοδοτήσει πώς φαντάζεται βραχυπρόθεσμα μια στρατηγική ε, σε περίπτωση ε, που κάνουν οι εξτρεμιστές ε, αυτό που ήδη έχουν εξαγγείλει, ότι θα πλημμυρίσουν τη Μεσόγειο με μετανάστες και πρόσφυγες. Και υπάρχουν χώρες της Μεσογείου που θα πληγούν ιδιαίτερα. Ποιος θέλει να λάβει το λόγο υπέρ αυτού του αιτήματο. κυρία Μέτσολα. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όντως, η κατάσταση ασφαλείας στη Λιβύη μας ανησυχεί πολύ Όλο και περισσότεροι άνθρωποι από διάφορες εθνικότητες, ακόμα και υπήκοοι των Ηνωμένων Πολιτειών, απάγονται από εκπροσώπους του Ισλαμικού κράτους. Επίσης βλέπουμε ότι προελάβει το Ισλαμικό κράτος σε διάφορες παραθαλάσσιες πόλεις της Λιβύης και βλέπουμε ότι κινδυνεύουν πάρα πολλοί άνθρωποι με εκτοπισμό, καθότι θέλουν με κάθε τρόπο να φύγουν από το καθεστώς αυτός τρόμου που ισχύει στην Λιβύη. Συνεχίζονται όμως και οι συζητήσεις στα Ηνωμένα Περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να γνωρίζουμε ποια θα είναι η δική της τακτική, πώς μπορεί να δραματίσει ένα σημαντικό ρόλο. Οι πολίτες μας ανησυχούν όλο και περισσότερο, ζητούν μία ανταπόκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά την κατάρριψη του Καντάφη, πολλέ χώρε, και ιδιαίτερα η Ιταλία δέχθηκαν πάρα πολλού μετανάστε. Κάνω λοιπόν έκκληση προ όλου να αφήσετε κατά μέρο οποιαδήποτε πολιτική προσέγγιση για το ζήτημα αυτό και να καταφέρουμε από κοινού να βρούμε μία λύση για την κρίση στη Λιβύη. Και α μην περιμένουμε να χαθούν πάλι πάρα πολλέ ζωέ. Α κάνουμε πρώτα μία συζήτηση εδώ πέρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Κατά ο κύριο Γκερέρο. Ευχαριστώ. Όχι, δεν είμαστε στην ουσία κατά, αλλά έχουμε μία εναλλακτική πρόταση. Δηλαδή, αντί να επικεντρωθούμε αποκλειστικά στις μεταναστευτικές ροές, καλό θα ήταν να μιλήσουμε για την κατάσταση της Λιβύης και τον κίνδυνο που δημιουργεί αυτή η αστάθη, η έλλειψη κυβέρνηση, η ακυβερνησία που επικρατεί στη Λιβύη και τι μπορούμε να κάνουμε για να συμβάλλουμε στη σταθεροποίηση της κοινωνίας και της ε, πραγματικότητας στη Λιβύη. Και στο πλαίσιο αυτό να εξετάσουμε και το θέμα της ροής των μεταναστών. Δηλαδή, να μιλήσουμε για τη Λιβύη και όχι μόνο και μόνο για τις ροές των μεταναστών που φτάνουν μέχρι τις ακτές μας. Κύριε Γκερέρο, θα πρέπει πρώτα να ψηφίσουμε την αρχική πρόταση. Γιατί η δική σας είναι μια εναλλακτική πρόταση, δεν είναι αντίθετη. Λοιπόν, πρώτα να ψηφίσουμε το αίτημα της κυρίας Χολμάγερ. Ή θέλετε το λόγο κυρία Χολμάγερ για να αποφαθείτε για το όσο είπε ο κύριος Γκερέρο για την πρότασή του. Κύριε Πρόεδρε, δεν θα μπορούσαμε να δούμε ένα κοινό τίτλο να πούμε πρώτα Λιβύη και μετά οι επιπτώσεις στη μετανάστευση κτλ. Και άλλα θέματα, τρομοκρατία, να είναι μια κοινή επικεφαλίδα. Λιβύη συν τα διάφορα θέματα. Κύριε Γκερέρο, ορίστε τώρα ανοίξαμε δουλειές. Μα αυτό σας είπα κι εγώ να γίνει μια γενική συζήτηση για την κατάσταση στη Λιβύη, τους πιθανούς κινδύνους που εγκυμονούν εκεί οι καταστάσεις και τι επιπτώσεις θα έχει αυτό στις μεταναστευτικές ροές. Κάπως έτσι θα μπορούσε να είναι η επικεφαλίδα. Λοιπόν, ο Πρόεδρος. Θα μπορούσαμε λοιπόν να συμφωνήσουμε να γράψουμε στην ημερήσια διάταξη δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αποσταθεροποιημένη κατάσταση στη Λιβύη και τις επιπτώσεις που απορρέουν από αυτή που συνδέονται. Κάπως έτσι. Ωραία. Ποιος συμφωνεί με την πρόταση αυτή του Προέδρου. Παρακαλώ ψήφιπε. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται λοιπόν ούτως. Ευχαριστώ πολύ. Ορίστηκε η διάταξη των εργασιών.